So, meine Damen und Herren. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι λοιπόν. Ακολουθούν επεξηγήσεις ψήφου. Zur Abstimmung und dabei beginnen wir mit Αρχίζουμε με κίνες τις επεξηγήσεις ψήφου που δεν μπόρεσαν να κατατεθούν την Τρίτη παρακαλώ. Μετά έχουμε τις επεξηγήσεις για τα χτεσινά, της Τετάρτη και μετά της Πέμπτης. Πρέπει να σα ενημερώσω ότι έχουμε πάρα πολλές αιτήσει για προφορικές ε, επεξηγήσεις ψήφου. Μέχρι τη μία μισή όμως θα κρατήσει συνεδρίαση και οι υπόλοιπε μπορούν να κατατεθούν γραπτός. Αρχίζουμε λοιπόν από την έκθεση του κυρίου Φέρμπερ για την αυτόματη ανταλλαγή προφοριών στη φορολογία την υποχρέωση αυτή. Η συνάδελφος Παλώμα Λόπερ ε, Μπερμέχο έχει ζητήσει, αλλά δεν τη βλέπω στην αίθουσα. Η Κριστίνα Μόρβαη, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Εγώ υποστήριξα τους νέους κανόνες που ήταν απαραίτητοι. Απαραίτητοι. Μετά την, υπό την ηγεσία του κ.